<clears throat> Dzień Κυρίες και κύριοι, σα εύχομαι καλώς ήρθατε. Κυρίσω την έναρξη λοιπόν της ε, συνόδου. Πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης αφορά τη συζήτηση, την κοινή συζήτηση όσον αφορά τον προπολογισμό